δεν πρέπει να εγκριθούν αυτέ οι διατάξει, δεν νομίζω ότι είναι καν λογικό σε όρου ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κράμερ και συγχαρητήρια για την πολύ καλή σα δουλειά. Η, συζη... η, ολοκληρώ... η συζήτηση που ολοκληρώθηκε, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στι 12 το μεσημέρι και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι πλέον και το τελευταίο τέτοια ώρα. Είναι η έκθεση της κυρίας Χάση σε σχέση με τη θέση υποχρεώσεων των φορών εκμετάλλευση που διαθέτουν ξυλία και προϊόντα ξυλία στην αγορά. Και ευχαριστώ και συγχαίρω την κυρία Χάση, η οποία ανέλαβε ε, στα μισά του δρόμου την έκθεση αυτή, γιατί η αρχική συγγετρία κυρία Λούκα παραιτήθηκε από την έδρα τη για να αναλάβει άλλα καθήκοντα στο Εθνικό τη Κοινοβούλιο. Η κυρία Χάση, λοιπόν, έχει το λόγο ω εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κυρία Λούκα και του διαπραγματευτέ από τι άλλε πολιτικέ ομάδε για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστούμε επίση και την ε, Ισπανία, η οποία, ε, την Ισπανική Προεδρία που διεξήγαγε τι διαπραγματεύσει σε επίπεδο Συμβουλίου, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που άλλαξαν σημαντικά και η Επιτροπή και το Συμβούλιο την αρχική του θέση για να ε, κλείσουμε τις αγορές μας ε, στην ε, παράνομα υλοτομημένη ξυλία. Αυτό δεν μπορούσε να έχει επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη και της πλειοψηφία του Κοινοβούλιο. Τώρα συμφωνήθηκε η σαφής απαγόρευση αυτών των προϊόντων και οι, οι, οι, λιανέμποροι θα πρέπει να αποδεικνύουν από πού ε, αγόρασαν την ξυλία, ποιος την πούλησε δηλαδή. Ε, αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση. Έτσι μπορούμε να δούμε την προέλευση του ξύλου που χρησιμοποιείται για παράδειγμα για την κατασκευή επίπλων. Δεν θέλαμε λοιπόν ε, η απαγόρευση να ισχύει μόνο για το πρωτοτμήμα της αλυσίδας. πρέπει να δούμε ε, και τι γίνεται στα υπόλοιπα τμήματα της αλυσίδας. Όλοι λοιπόν αναλαμβάνουν τις ευθύνε τους και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μην ε, πολλούν παράνομα ελαττωμένη ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει τις σοβαρές παραβάσεις στο θέμα της ε, ε, παράνομης, ε, παράνομα ελαττωμένης ξυλίας να θεωρούνται ως, ως πραγματικά ποινικά αδικήματα. Και κοιτάξτε, όσον αφορά τον κίνδυνο και τον αμεληταίο κίνδυνο φαίνεται ότι είναι, υπάρχει ένα σχεδόν μηδενικός ε, ε, κίνδυνο όσον αφορά για παράδειγμα ε, τους ε, ε, ε ορισμένους μικροοργανισμούς ε, στα, στα τρόφιμα κτλ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά στη συναφή νομοθεσία θεωρεί ως αμεληταίο κίνδυνο τον κίνδυνο που πρακτικά είναι μηδενικός. Και θα ήθελα να αναφέρω το γεγονό ότι ε, επειδή ορισμένα προϊόντα δεν συμπεριλαμβάνονται στην νομοθεσία, μπορεί να δημιουργηθούν παραθυράκια. Όσον αφορά δηλαδή ε, το έντυπο υλικό, για παράδειγμα, ε, το χαρτί ε, που παράγεται στην Τουρκία και αλλού, στην Κίνα και αλλού. Κοιτάξτε, το 20% των εκπομπών οφείλονται στην παράνομη υλοτόμηση, ενώ ταυτόχρονα καταστρέφεται και η βιοπικιλότητα. Λόγω της παράνομης υλοτομίας, Ε, δεν μπορεί να γίνεται έρευνα ε, για ορισμένα φάρμακα, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρόνια ε, αγωνίζεται κατά της παρανομη υλοτόμησης, αλλά ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές. Παρά τα λόγια λοιπόν, εμείς συμβάλλουμε στην ουσία στην καταστροφή των δασών. Το γεγονό λοιπόν ότι τώρα την απαγορεύουμε πραγματικά την ε, παράνομη υλοτόμηση, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα σε παγκόσμιο επίπεδο και δείχνουμε το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις, ε, μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα ε, για την επίλυση των, των, προβλημάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Δίνουμε λοιπόν το παράδειγμα με αυτή την νομοθεσία. και συμβάλλουμε ε, στην, στον τερματισμό αυτού του φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστούμε και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ποτότσνικ για να τοποθετηθεί εξ ονόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, Πρόεδρε, εξωτμή. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερω τι δύο εισηγήτριε, την κυρία Καρολάιν Λούκα και την κυρία Χάση, καθώς και τους σκιώδεις ηγητές για την ε, συνεργασία τους, ε, τη βούληση για συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή που οδήγησε στο συμβιβασμό που έχουμε μπροστά μας. Τα δάση έχουν ζωτική σημασία και για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και για την προστασία από την κλιματική αλλαγή και την ε, προστασία των υδάτων στον πλανήτη μας. Δεν είναι πουθενά σαφέστερη εικόνα της πληρότητας της οικολογικής ισορροπίας όσο στα δάση. Γι' αυτό λοιπόν και η οικονομική αλλά και η κοινωνική αξία των δασών είναι τεράστια. Εγώ από τη δική μου την πατρίδα, όπου καλύπτουν περίπου 60% της επικράτειας τα δάση, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη σημασία τους. Είναι σε πολλές χώρες τα δάση όχι μόνο πηγή εργασίας, αλλά και ε, φαρμάκων, ειδών τροφής, διατροφής, στέγης Τεράστιες σημασία λοιπόν για τι κοινωνίε μα τα δάση και γι' αυτό θα πρέπει η ψηφοφορία με τη δεύτερη ίσως ανάγνωση να αποτελέσει ένα σαφέ μήνυμα για ολόκληρο τον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται την λαθρέα υλοτόμηση και τα προϊόντα αυτή. Το... Η μεγάλη πρόκληση είναι πώ διαγιγνώσκεται ότι ένα είδο ξυλία, προϊόν ξυλία προέρχεται από λαθρέα υλοτόμηση. Εδώ καλύπτεται μόνο το είδο ξυλία το οποίο εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια τι προσπάθειέ τη ε, για τα, με τα κράτη εκείνα τα οποία επιδιώκουν μια καλύτερη διαχείριση των δασών του, τα τρίτα κράτη. Πιστεύω ότι πολύ σωστά η έκθεση αυτή αναγνωρίζει τη σημασία των συμφωνιών που μπορεί να συνάπτουν τα τρίτα κράτη με την Ευρωπαϊκή Ένωση το να θεωρηθεί ότι με τη συμφωνία αποτελεί επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες δασών δεν ευσταθεί κατά την απόψή μου γιατί προσφέρεται επαρκή ευελιξία από το κείμενο της ε, οδηγίας και θα ήθελα να πω ότι η έκθεση που έχετε ενώπιον σας ε, αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδο και ελπίζω να την υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στους ομιλητές εξ των ε, κοινοβουλευτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα για δύο λεπτά το λόγο ο κύριος Φιέλνερ, μιλώντας εξ ονόματο του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστώ θερμά την κυρία Χάση. Είναι καιρό που μα απασχολεί αυτό το νομοθέτημα. Είναι καιρό που λέμε ότι χρειαζόμαστε καλή συνεργασία στο θέμα της ε, ε, εκμετάλλευση των δασών μας. Έχω λοιπόν τα εξής ερωτήματα. Το ξύλο είναι ένα καταπληκτικό, ανανεώσιμο, αξιοποιήσιμο και ε, α, καλής ποιότητας υλικό. Όμως βλέπω δυστυχώς εδώ ότι η νομοθεσία μπορεί να επιβάλλει ε, δυσμενή μεταχείριση του ξύλου και των προϊόντων ξυλίας έτσι ώστε τελικά να προτιμά κανείς την, ε, τα, προϊόντα από, τα αντίστοιχα προϊόντα από μέταλλο ή πλαστικό. Ευτυχώς όμως αυτό θα το αποφύγουμε ελπίζω. Επίσης, πρέπει να φροντίσουμε όταν έχουμε να κάνουμε με προϊόντα μεταποιημένα, προϊόντα ξυλίας μεταποιημένα, να είμαστε θέση να ε, ανοιχνεύσουμε την προέλευσή τους. Να ξέρουμε εάν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από λαθρέα υλοτόμηση. Και τρίτον, η νομοθεσία θα πρέπει να εισάγεται χωρίς όμως να αποτελεί μη δασμολογικό φραγμό στην εισαγωγή των προϊόντων αυτών από τρίτα κράτη. Θα πρέπει να σε θέση να εισάγουμε αλλά και να εξάγουμε τα προϊόντα ξυλίας εφόσον έχουν τηρηθεί οι κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της. Πιστεύω ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό έργο και κλείνοντας θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους και να τους υπενθυμίσω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη λαθρέα ελοτόμηση και ταυτόχρονα θα πρέπει να πατάξουμε την νομοθεσία αυτή, τη διαφθορά και την εγκληματικότητα που αναπτύσσεται πέρι τη λαθρέα αυτή ελοτόμηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φιέλλερ. Το λόγο έχει ο κύριος Αρσένης για δύο λεπτά εκ μέρους των Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτροπέ Ποτότσνικ είναι πραγματικά μια συγκινητική στιγμή, μια ιστορική στιγμή και η σημερινή συζήτηση και η αυριανή ψηφοφορία. Ε, πραγματικά βλέπω πολλούς φίλους που δώσαμε έναν ε, σκληρό αγώνα μαζί και καταφέραμε να φέρουμε ε, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο αρκετά κοντά στις αρχικές θέσεις του Κοινοβουλίου, αρκετά να έχουμε μπροστά μας μια νομοθεσία ε, που προστατεύει και τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Μέχρι σήμερα η ένας Ευρωπαίος πολίτης όταν αγόραζε ξυλία και προϊόντα ξυλίας δεν μπορούσε να γνωρίζει αν είναι νόμιμη ή παράνομη. Αν αγοράζοντας επιδοτεί αιματηρούς εμφύλους πολέμους ε, που γίνονται με, χρηματοδοτούνται μέσα από την παράνομη λοτόμηση ή και την κλιματική αλλαγή μέσα από την αποδάσωση αυτή τη στιγμή με αυτή την νομοθεσία ε, και την προσπάθεια του κοινοβουλίου καταφέραμε να συμφωνήσει και το συμβούλιο στο αυτονόητο το η παράνομη ξυλία να θεωρείται παράνομη και στην ευρώπη. καταφέραμε επίσης η όρη, η έγκριση η εξουσιοδότηση των φορέων που θα επιβλέπουν ε, την, ε, τα συστήματα αξιολόγηση της νόμιμης ξυλίας που θα δίνουν δηλαδή την έγκριση ε, στα προϊόντα ξυλίας ε, να γίνεται ο έλεγχος αυτός να γίνεται κεντρικά μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταφέραμε όταν θα εξετάζει ο κάθε φορέας αν μια ξυλία είναι νόμιμη να συμπεριλαμβάνει και νομοθεσία που αφορά τη βιοπικιλότητα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά πολλά σημεία, υπάρχουν δύο κεντρικά σημεία τα οποία το Συμβούλιο ε, δεν δέχτηκε και γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Δεν δέχτηκε το Συμβούλιο, ε, κατά τη γνώμη μου, κάτι αυτονόητο, το ότι θα έπρεπε αυτή, αυτό το, το παράπτωμα πλέον, το να εισάγει κανείς ε, για πρώτη φορά παρά, παράνομη ξυλία στην ευρωπαϊκή αγορά και προϊόντα ξυλίας να σωματωθεί στην οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα είναι κάτι εντελώ παράλογο όπω δεν ε, εισάγει και διατηρεί την έννοια ε, του αμεληταίου κινδύνου ε, ανοίγοντα ένα παράθυρο για μερικέ δραστηριότητε να μην χρειαστεί να ακολουθήσουν διαδικασίε που προβλέπει η νομοθεσία. όμω αυτή η νομοθεσία προστατεύει τον ευρωπαίο πολίτη προστατεύει τον ευρωπαίο παραγωγό από τον αθέμητο ανταγωνισμό και από χαμηλές τιμές που έχει μοιραία η παράνομη ξυλία και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και συνεργάτες που έχουν δουλέψει για αυτό το θέμα όπως είναι ο Αλέξανδρος ο και όλο το γραφείο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Εξ ονόματος των Φιλελευθέρων για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Γκερμπραντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής. Όχι μόνο γιατί κέρδισε η Ολλανδία εναντίον τη Ουρουάη στους ημιτελικού, αλλά και γιατί περνάει ένα σαφές μήνυμα ε, προς τον υπόλοιπο κόσμο με αυτό το κείμενο. 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αποφάσισαν ότι δεν θέλουν ξύλο ή προϊόντα ξύλου που υλοτομούνται παράνομα. Και όσοι προσπαθούν, προσπαθήσουν να αγοράσουν τέτοιο ξύλο θα υποστούν κυρώσει. Είναι σαφέ αυτό το μήνυμα. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία του. Η αποψήλωση των δασών παραμένει παγκόσμιο πρόβλημα τεράστια εμβέλεια. Εμεί, οι καταναλωτέ Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μία δύναμη που έχει η πυρός μας, την ε, δυνατότητα κατανάλωσης για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα καταφέραμε. Το Συμβούλιο λοιπόν θέλει να αποθαρρύνει την ε, παρανομιλοτόμηση, ενώ εμείς θέλουμε να απαγορεύσουμε την παράνομη υλοτόμηση. Ε, δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοια εισαγωγή τέτοιου ξύλου. Αυτό είναι νίκη τη ε, δημοκρατία. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Ισπανική Προεδρία και τη Βελική Προεδρία, η οποία δεν είναι παρούσα βέβαια, για αυτή τη νίκη. Ε, και ελπίζω τελικά να καταφέρουμε να έχουμε μια πλειοψηφία στο Συμβούλιο εναντίον της απαγόρευσης. Θα ήθελα ε, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου να παγρυπνήσουν τόσο ώστε να εφαρμοστεί αυτή η νέα νομοθεσία. Γιατί αυτό είναι το κλειδί τη επιτυχία τη νέα νομοθεσία. Αν δεν την εφαρμόσουμε αποτελεσματικά, θα παραμείνει γράμμα κενό περιεχομένου. Συμπερασματικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάση, καθώ και την κυρία Λούκα, για τη θαυμάσια δουλειά και τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση και του κοιόδη εισηγητέ. Νομίζω ότι δώσαμε το παράδειγμα. Δείξαμε πώς εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να ασκήσουμε το δημοκρατικό μας βάρος ε, και κύρος ε, υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο η κυρία Γκέρλινγκ εξ ονόματος της ομάδας ECR. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ ε, ε να συγχαρώ τον συγκητή γιατί πραγματικά και την συγκήτρια γιατί πραγματικά ε, υπήρξε αίσιο τέλος και χαίρομαι και εγώ που συμμετείχα σε αυτές τις ε, ε, συζητήσεις. Από τη μια μεριά προστατεύονται τα δάση και η βιοπικιλότητα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και απαραίτητη ευελιξία για να μην ε, επιβληθεί υπερβολικό βάρος στους νόμιμους και ειλικρινείς εμπόρους. Είναι λοιπόν δυνατό να υπάρξει τέτοια συμφωνία αν όλοι συνεργαστούμε από κοινού. Θα ήθελα να τονίσω ε, ένα σημείο ε, και και, για μένα είναι ευτυχή συγκυρία που ασχολήθηκα με το ζήτημα αυτό. Μιλώ ε, για μια ε, παράπλευρη επίπτωση. Η Αναφέρομαι στη συνειδητοποίηση των ε, πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε συνειδητοποίηση και, και μια δημόσια συζήτηση. για μένα, που είμαι νέο μέλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν, η συνειδητοποίηση του κοινού ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πολίτες εντυπωσιάστηκαν από την ε, συμβολή του Κοινοβουλίου, το οποίο όφησε την νομοθεσία προς την κατεύθυνση που και το κοινό επιθυμεί. Ε, ευχαριστώ λοιπόν όλους και ήταν για μένα πραγματικά μάθημα που συνεργάστηκα με την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε. Δυόμιση λεπτά τώρα έχει το λόγο η κυρία Ματίας εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες για τη θαυμάσια δουλειά τους. Νομίζουμε, νομίζω ότι η παρο, παράνομη υλοτόμηση είναι μεγάλο πρόβλημα για το παγκόσμιο περιβάλλον. Αποψηλώνονται εκατομμύρια εκταρίων και αυτό είναι μεγάλη απειλή για την βιοπικιλότητα. Η αποψήλωση των δασών η αποδάσωση είναι κάτι το οποίο έχει αρνητική επίπτωση. Κανένας δεν, το, δεν αρνείται αυτό το πρόβλημα. Ε, επίσης ε, εξηγεί έτσι και κάποια ακραία κλιματικά φαινόμενα που έχουμε σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Είναι μεγάλος κίνδυνος λοιπόν για όλο τον πλανήτη μας αυτός. Φυσικά ε, δεν το υφιστάμεθα αυτό το πρόβλημα όλοι στον ίδιο βαθμό. Οι κοινότητες οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από τα δάση για την επιβίωσή τους είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο. Είναι σαφές επίσης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κατανομής των φυσικών πόρων και ένα πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πληθυσμούς αυτούς που ζουν από τα δάση. Η θέση σε εμπορία παράνομου ξύλου αντιπροσωπεύει το 20% του συνόλου του ξύλου. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιλύσουμε το πρόβλημα και για τις χώρες παραγωγούς και για τις χώρες που καταναλώνουν το ξύλο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τρόπο βιώσιμο αυτό το φυσικό υλικό που είναι το ξύλο. Δεν έχει νόημα να, να μασάμε ωραία και μεγαλόστομα λόγια, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Η έκθεση αυτή μας επιτρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, ένα αποφασιστικό βήμα για την διαχείριση ε, του ξύλου. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, πρέπει να είμαστε και αποτελεσματικοί. Χρειαζόμαστε κυρώσει, κυρώσεις αποτρεπτικές, αποτελεσματικές καταρχάς πρόστιμα και από την άλλη, εάν υπάρχει επανάληψη του λάθους, θα πρέπει να υπάρξει κατάσχεση του εν ξύλου και άρση των αδειών για τη θέση σε εμπορία αυτού του ξύλου. Εκείνοι που θέτουν σε εμπορία φυσικούς σπόρους θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι απέναντι στην κοινωνία. Επομένως, εκείνοι οι οποίοι θέτουν ε, ξύλο ε, στην ευρωπαϊκή αγορά για πρώτη φορά θα πρέπει να σέβονται τα μέτρα που είναι ενισχύ και να λογοδοτούν σε όλα τα θέματα που φορούν την προέλευση του ξύλου. Οι πληθυσμοί, οι κοινωνίες μας θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ε, στην ενημέρωση. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιος δεν σέβεται αυτούς τους κανόνες. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ροσβάχα, εκ μέρου τη ομάδα τη Ευρώπη των Ελευθεριών και τη Δημοκρατία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. ιδιαίτερω για την προσπάθεια που ανέλαβε η κυρία Χάση στα μισά του δρόμου ανέλαβε μια πολύ περίπλοκη νομοθεσία. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ε, τα δάση μας από την παράνομη λοτόμηση, να διαφυλάξουμε τη βιοποικιλότητά μας και να προστατεύσουμε την αγορά μας από τα μεταποιημένα προϊόντα που έχουν παράνομα υλοτομηθεί, προέρχονται από ξυλία παράνομα υλοτομημένη έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν κάποιο προϊόν έχει παραχθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθείται από ένα πιστοποιητικό ε, υλοτόμ, νόμιμης υλοτόμησης και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να ελεγχθεί η προέλευσή του. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με ξυλία και πάνω απ' όλα με προϊόντα μεταποιημένα που προέρχονται από τρίτες χώρες, παραδείγματι ε, έπιπλα, από MDF ε, ή προϊόντα μεταποιημένης ξυλίας, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι οι δραστηριότητες ε, της μεταποίησης να δεφυλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία και τώρα μπορούμε να περάσουμε σε επιμέρου ομιλητέ. Πρώτα απ' όλα για 1,5 λεπτό η κυρία Πιετικάινεν. Σα ευχαριστώ. Πράγματι έχουμε ένα βήμα προς την χρήση, ορθολογική χρήση των πόρων αυτών ε, και ανάληψη ε, ευθυνών σε παγκόσμιο επίπεδο, προστασία βιοποικιλότητας και βελτίωση του επίπεδου ζωής των, ε, των πολιτών. Μπορούμε να δείξουμε τον τρόπο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτελεσματική ως, σε διεθνές επίπεδο ακολουθώντας αυτή την νομοθεσία, η οποία συμφωνεί και με τα οικολογικά πρότυπα. Το αποτέλεσμα σαφώς είναι καλύτερο από ε, το, το αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο παρά τα μειονεκτήματα που υπάρχουν. Και θα ήθελα να πω και εγώ ότι ε, βεβαίω ένα από τα μειονεκτήματα είναι το γεγονός ότι ε, δεν προβλέπονται κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και επίση ε, ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία που αναφέρεται στα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Δηλαδή ότι η παράνομη υλοτόμηση δεν συμπεριλαμβάνεται ε, στο συγκεκριμένο σημείο. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλει προτάσει και προ την κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή. Ε, Επίση, όπω ε, όπως ακούσαμε, και το έντυπο υλικό και το χαρτί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Ευχαριστούμε. Τώρα δυόμιση λεπτά έχει το λόγο η κυρία Λίντα Μακάβαν. Πρόεδρε. Περασμένη ώρα, συνάδελφοι. αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικέ προφορίες ε, τη ε, εβδομάδα που διανύουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό βλέπω και από το ταχυδρομείο που λαμβάνω, από τα πολυάριθμα γράμματα και 125.000 υπογραφές σε μια ε, διαδικτυακή αναφορά που μας καλεί να υποστηρίξουμε τις προτάσεις αυτές με την αυριανή ψηφοφορία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε, νομίζω, ότι έχει τεράστια σημασία αυτή η νομοθεσία και για τα εκατοντάδε εκατομμυρίων πολιτών των φτωχότερων χωρών που υποφέρουν από την λαθρέα υλοτόμηση. 100.000 ήταν τα δέντρα τα οποία ε, υλοτομήθηκαν παράνομα στην Μαδαγασκάρη πέρυσι. Τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας και βέβαια εγκληματικότητα συναφής με αυτή. Η Λιβερία, παραδείγματι, 250.000 ανθρώπους κατάφερε να σκοτώσει εκμεταλλευόμενοι τα έσοδα της παράνομης ξυλίας της. Το ίδιο και στην Καμπότζη, στη δεκαετία του 90. Έτσι λοιπόν το Global Witness, η οργάνωση αυτή φαίνεται έχει υπολογίσει ότι το καθεστώς της Κίνας εκμεταλλεύεται ε, την, ε, εκμεταλλεύεται την ξυλία της Βυρμανίας και τα αντίστοιχα της προσφέρει προστασία στο παράνομο καθεστώς της. Η Human Rights Watch λέει ότι 2 δισεκατομμύρια δολάρια από ε, έσοδα φορολογικά της Ινδονησίας έχουν απολεστεί λόγω της παράνομης υλοτόμησης. Θα είχαν σωθεί πολλές ανθρώπινες ζωές, εκατοντάδες χιλιάδων Ινδονησίων θα είχαν μια αξιοπρεπή ατροφαρμακευτική περίθαλψη αν υπήρχαν αυτά τα φορολογικά έσοδα. Και ναι μεν δεν είναι τέλεια η, η νομοθεσία αυτή που έχουμε να ψηφίσουμε αύριο, αλλά είναι πολύ καλύτερη από την λεγόμενη αρχή της διοντολογικής προσαρμογής, της δέουσας ε, προσοχής και της εθελοντικής προσαρμογής. Είναι πολύ καλύτερη, ευχαριστώ την Ισπανική Προεδρία για την στήριξή της και ευχαριστώ και τον Υφυπουργό της Βρετανίας για την υποστήριξη μας προς σε επίπεδο Συμβουλίου για μια πιο φιλόδοξη νομοθεσία. Είναι καλή δουλειά λοιπόν που έχουμε κάνει όλοι μαζί και οι σκιώδεις και η συγγήτρια. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε τις πιέσεις και να αφυπνίσουμε τους συμπολίτε μας την κοινή γνώμη για μια καλή υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της πολύ καλής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει 1,5 λεπτό ο κύριος Κρίς Ντέιβις. Ε, καταστρέφονται τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, μερικές φορές με την υποστήριξη των κυβερνήσεων, μέσω παράνομων δραστηριοτήτων συχνά. Ε, και μιλάμε για δραστηριότητες που γεννούν πάρα πολύ χρήμα που διαφθείρει τις κυβερνήσεις ε, και δυσκολεύει πολύ την εφαρμογή της νομοθεσίας. Πριν από πέντε χρόνια μίλησα με τον τότε επίτροπο, τον Λουί Μισελ, και του είπαμε χρειαζόμαστε τέτοια μέτρα. Εκείνος έτεινε δίκο νους ε, αλλά οι δικηγόροι του είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα, μπορούσαν, δεν θα μπορούσε να γίνει. Και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Επίτροπε. Εάν οι δικηγόροι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλάξτε του δικηγόρου. Ε, έχουμε την απόδειξη ότι μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η οδηγία λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν κάποια καθεστώτα εφαρμογής που είναι αποτελεσματικά, αποτρεπτικά και αναλογικά. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Τι λέει η Σλοβενία. Ποια είναι η ποινή για την παράνομα υλοτομημένη ξυλία. Θα είναι λέει 10 ε, χρόνια φυλακής. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο λέει «Α, τίποτα, ε, μία επίπληξη ας πούμε». Δεν, είναι, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε έτσι με τελείως διαφορετικό τρόπο αυτή την νομοθεσία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, δημοσιοποιούν τις ε, λεπτομέρειες των κυρώσεων που επιβάλλουν, ούτως ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η νομοθεσία. Θα πρέπει να ονοματίζουν, να στυλιτεύουν με πρωτοφανή τρόπο. Κύριε Επίτροπε, ε, αποτελεσματικά, αποτρεπτικά και αναλογικά. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα λόγια. Θέλω αυτά τα λόγια να έχουν και ουσία από πίσω και εσείς να είστε το Επίτροπος που το εξασφαλίσει αυτό. το για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παράγουμε καλή νομοθεσία σήμερα. Καλή και χρήσιμη για την αποφυγή της κυκλοφορίας παράνομων προϊόντων υλοδόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όπως και για κάθε νομοθέτημα δεν πρέπει να περιλαμβάνει αυτά που θα θέλαμε να περιλαμβάνει, αλλά να κοιτάμε αυτά που γράφουμε, αυτά που προδιαγράφουμε από την νομοθεσία να είναι και εφαρμόσιμα και να εφαρμόζονται πράγματι. Με το συμβασμό λοιπόν, το πρώτο σημείο, η επαγρύπνηση κατά την ε, θέση σε κυκλοφορία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και εφαρμογή κατά την θέση σε κυκλοφορία μέσα στην Ευρώπη προϊόντων αυτών. Δεν είναι δυνατόν όμως από την στιγμή που θα μπαίνει ένα προϊόν ξυλίας μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθείται από μία σειρά εγγράφων και προστοποιητικών που θα καθυστερούν την ε, μεταποίησή του και την αξιοποίησή του στην αγορά. Είπε και η κυρία Χάση νωρίτερα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία πολιτική αμεληταίου κινδύνου, μάλλον μηδενικό κίνδυνο δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί, μπορεί, γιατί το μόνο που θα παραγάγει είναι επιπλέον γραφειοκρατία και άρα περισσότεροι κίνδυνη. Πρέπει να έχουμε μια, μια νομοθεσία εφικτή και αποτελεσματική, πραγματοποιήσιμη δηλαδή, όπω αυτή που έχουμε τώρα, την οποία ελπίζω θα στηρίξει αύριο η πλειοψηφία των συναδέλφων. Ευχαριστώ για ένα λεπτό τώρα η κυρία Μάνερ. Πρόεδρε. Πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα στη λαθρή ολοτόμηση. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, πιστεύω. Όμως δεν υποστηρίζω πλήρως τον ε, συμβασμό. Το ζήτημα της ευθύνης, παραδείγματι, της παρακολούθησης κάθε σημείου της αλυσίδας της κυκλοφορίας του προϊόντος, μάλλον θα επιβαρύνει το γραφειοκρατικό άχθος για τις επιχειρήσεις και βέβαια δεν πρέπει να είναι αυτό ο στόχο που επιδιώκουμε. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κατά την υλοποίησή της η νομοθεσία αυτή θα έχει μέτρα πιστοποίησης, διατάξεις σχετικέ με την πιστοποίηση των προϊόντων, εφικτά και όχι απαιτήσει υπερβολικές ή αλληλεπικαλυπτόμενες. Επίσης δεν πρέπει το ξύλο να έχει δυσμενέστερη μεταχείριση από ό,τι άλλα προϊόντα. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ε, ομιλητής, ο κύριος ε, Χάγκλουντ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς. Ένα τόσο σημαντικό θέμα θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε. Το είπε και ο κύριος Μάνερ νωρίτερα. Είναι λυπηρό το ότι μερικές φορές λησμονούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σημαντική παραγωγή ξύλου, με ένα πολύ σημαντικό κλάδο, τον κλάδο της φιλετομίας, της αστικής παραγωγής, που, είναι, που έχει μεγάλη σημασία οικονομική και κοινωνική στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Χάση και όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν στην νέα αυτή πολύ καλή νομοθετική πρόταση. Πρόταση που βελτιώνει τις προτάσεις της Επιτροπής. Ο βεσμός είναι καλός πιστεύω και εξασφαλίζει την ε, απαγόρευση της ε, παράνομης υλοτομίας χωρίς όμως να πλήττεται η θεμητή, νόμιμη και οργανωμένη υλοτομήση. Ευχαριστούμε κύριε Χάγκλουν. Τελειώσαμε λοιπόν με, το, με τους ομιλητές στο Catch the Eye. Με τους ομιλητές μάλλον και περνάμε τώρα ε, στο, στο Catch the Eye ε, όπου έχουμε τρεις ομιλητές, τρεις συναδέλφους που έχουν ζήσει το λόγο και πρώτα απ' όλα η κυρία Αντωνέσκου. Ένα λεπτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το εμπόριο ξυλίας ε, της ε, ε, ε, παράνομης ξυλίας μειώνει την τιμή του ξύλου και υποβαθμίζει τα δάση. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται η συγκεκριμένη νομοθεσία. Η νομοθεσία αυτή εισάγει αυτό το σύστημα της δέουσας προσοχής και προβλέπει εποπτεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συστήματα λοιπόν αυτά θα προβλέπουν τον έλεγχο της ξυλίας που τίθεται στην αγορά. Βεβαίως η λύση που προτείνεται δεν είναι τέλεια, διότι ακόμα και το σύστημα αυτό είναι ευάλωτο και μπορεί να παρακαμφθεί. Γι' αυτό στι ε, συζητήσει στην αρμόδια επιτροπή πρότεινα μία τροπολογία λέγοντα ότι θα, ε, τα υποπτικά όργανα θα χάνουν τη διαπίστευσή του εάν ε, τελικά δεν χρησιμοποιείται ένα σύστημα δέουσης προσοχής. Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προ την κατεύθυνση της απαγόρευση παράνομης, παράνομα αλλά απαιτούνται και άλλα συστήματα. Ευχαριστούμε, λέει ο επόμενη ομιλήτρια. Το 2010, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είναι το έτος της βιοπικιλότητας και αυτό σημαίνει πολύ σημαντικέ ε, μέτρα σημαντικά για την προστασία της βιοπικιλότητας και, τη, και του περιβάλλοντος πρέπει να εισαχθούν. Όπως αυτό εδώ το νομοθέτημα για την, για την απαγόρευση της παρανόμης υλοτόμησης που αποτελεί ένα από τους κύριους παράγοντες αποψήλωσης των δασών από παράνομες ε, πηγές ξυλίας έχουμε περίπου 40% της ξυλίας παγκοσμίως αυτή τη στιγμή και 20% των ε, δασών που χάνονται στην, ε, στην θα μπορούσαν να έχουν απορροφήσει τεράστια ποσοστά διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν η απαγόρευση θέση τέτοιων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη και στέκεται υπεύθυνα κατά της παράνομης υλοτόμησης. Πρόεδρος Διακόπτη. Ευχαριστώ και τελειώνουμε με τον κύριο Πάσκα. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώνεται με την έκθεση Λούκας και Χάση είναι πάρα πολύ σωστή. Πρέπει να την υποστηρίξουμε, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καταπίνουμε την απροθυμία κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δεν θέλουν να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την παράνομη λοτόμηση και που δεν θέλουν ε, την εφαρμογή ε, κυρώσεων εναντίον αυτής της δραστηριότητας. Πάντως, Εξετάζοντας αυτή την νομοθεσία, τελικά ε, δεν ξέρουμε γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ε, είναι η απροθυμία των κυβερνήσεων, είναι η, το πείσμα κάποιων μαφιών. Ευχαριστούμε κύριε Πάστα. Τελειώσαμε με τους ομιλητές που πήραν το λόγο με διάφορη ιδιότητα ο καθένας και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Επιτρόπο κύριο Ποτότσινικ για να ε, απαντήσει ε, στα τα ερωτήματα και στις παρεμβάσεις και να κλείσει τη ζήτηση. Επίτροπο, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, έχει περάσει η ώρα και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Αυτό όμως ε, δεν σημαίνει ότι αποδίδω ε, μικρότερη σημασία στο ζήτημα, αλλά επειδή υπάρχει υψηλό βαθμό συνένεση στην αίθουσα. Κοιτάξτε, τα δάση βρίσκονται στο επίκεντρο του αγώνα για την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή και για την ε, προστασία τη βιοπικιλότητα. Μαζί με την πρόσφατη νομοθεσία για την παράνομη, ε, αδήλωτη και λαθρέα αλία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουμε ότι διαθέτουμε πλέον τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε την παρανομία σε δύο από τις, ε, από, τις βασικές από, δύο από τους βασικούς φυσικούς πόρους, αλία και την, δασοκο, και δασοκομεία. Και ταυτόχρονα που αποτελούν και μέσο για την καταπολέμηση της στόχιας. Ο, η, βεβαίως η νομοθεσία αυτή και η επιπτώση θα εξαρτηθεί από την πραγματική συμμόρφωση και η πρόκληση αυτή δεν έχει εξεπεραστεί. Αλλά μπορούμε από σήμερα να, να αρχίσουμε να βλέπουμε το γεγονός ότι ε, να, να βλέπουμε τα αποτελέσματα του γεγονότος ότι ε, υπήρξε μια συμφωνία σε αυτό το δύσκολο θέμα. Πραγματικά λοιπόν βρισκόμαστε απέναντι ε, σε μια ε, σωστή πρόταση και περιμένουμε ανυπομονησία να να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και σε επίπεδο διαδικασίας συμμόρφωσης με την οδηγία. Ευχαριστούμε κύριε Ποτόνι και σας ευχαριστώ και γιατί ήσασταν σύντομος και ε, συγκεκριμένος και περιεκτικός στην παρέμβασή σας και τελειώνει η σημερινή συζήτηση με την παρέμβαση της ε, εισηγητρίας της ε, κυρίας Χάση την οποία βεβαίω θα πρέπει να συγχαρούμε ε, και εκ μέρους του Προεδρείου, όπως άλλωστε έκαναν και όλοι οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο. Κυρία Χάση, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους σας, όλους όσους μιλήσατε τόσο αργά στη σημερινή συνεδρίαση. Και εγώ είχα εμπλακεί στην κατάσταση που περιέγραψε ο Chris Davis ε, στα πλαίσια της Επιτροπής Ανάπτυξης, όπου τότε Επίτροπος θεωρούσε ότι δεν ήταν δυνατή να προωθωθεί μια τέτοια νομοθεσία, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με υποστήριξαν ε, και μίλησαν για τα μειονεκτήματα της ε, παράνομης ξυλίας. Για όσους ανησυχούν για την επιπλέον γραφειοκρατία λόγω του νομοθετήματος αυτού, ε, θέλω να σας πω ότι δεν στοχεύουμε στο να καλύψουμε αυτούς που θέτουν για πρώτη φορά το ξύλο στην αγορά. Ε, δεν είναι σωστό μόνο για αυτούς, ε, αυτούς να τους βαραίνει ο πελεκής γραφειοκρατίας και τους υπόλοιπους όχι. Θα πρέπει όλοι να καλύπτονται. Και όλοι να, πληρούν, να πληρώνουν, να σέβονται τους κανόνες. Χαίρομαι που πολλές εταιρείες ε, υποστήριξαν την απαγόρευση της ε, παράνομης υλοτόμησης. Παραδείγματο χάρη στην τομέα του επίπλου και στην τομέα της συσκευασία. Πολλές εταιρείε μίλησαν υπέρ της απαγόρευσης. Ε, πολλά συνδικάτα επίσημα υποστήριξαν και είπαν ότι δημιουργείται ανταγωνιστικό μειονέκτημα ε, για αυτούς λόγω της ύπαρξης της παράνομης ξυλίας. Επομένως, τα κείμενα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν με το σωστό τρόπο και θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις από τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να μην υπάρχουν καθόλου καταχρήσεις του συστήματος. Σας ευχαριστώ κυρία Χάση. Με την παρέμβασή σα, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία, όπω είπαμε, θα γίνει αύριο το μεσημέρι στι 12 η ώρα. Συναδελφοί, η επόμενη ε, συνεδρίαση θα γίνει στις 7 Ιουλίου.